Now we are in an open session of this committee meeting. Our first item is item 10 on the protocol. Item 11, sorry. Αγαπητοί συνάδελφοι, ξεκινάει η δημόσια συνεδρία. Πρώτο σημείο, το σημείο 11. Διαδικασία έγκρισης συμφωνίες μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Δημοκρατία Αγίου Μαρίνου για προσαρμογή των εφιστάμενων συμφωνιών λόγω της προσχώρησης της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό βέβαια το απαιτεί ο ΠΟΕ, ξέρετε, οι υποχρώσεις μας δηλαδή απέναντι στον ΠΟΕ. Συγητής είναι υποφαινόμενος και δεν έχει αντιρρήσεις. Άρα μπορούμε να δώσουμε την έγκρισή μας στη συμφωνία αυτή που είναι κάτι που πρέπει να γίνει και με όλες τις χώρες, σε σχέση με όλες τις χώρες που έχουμε, όχι μόνο την Ελληνική Ένωση αλλά και συμφωνίες. Γιατί η υποσχώρηση της Κροατίας σημαίνει ότι η Κροατία πρέπει να για την Κροατία να ισχύουν ότι ισχύει για τους υπόλοιπους σε ό,τι αφορά τη σχέση με τις άλλες χώρες. uh, uh... Υπάρχει ατήρηση της ουσίας, ρωτώ τα άλλα μέλη της Επιτροπής. η ΕΕΔ που είναι υπεύθυνη για αυτό το φάκελο έχει να πει κάτι. Κανένα σχόλιο. Συμφωνείτε, λέει ο πρόεδρος. Δεν έχετε αντίρρηση, μάλιστα. Ναι, το σημειώνουμε. Ωραία. Επόμενο. Σημείο 12. Κατάσταση πρόοδο να τη Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών Ευρωπαϊκή Ένωση Βιετνάμ για τις διαπραγματεύσεις πρόκειται βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, θα εξετάσουμε τις τροπολογίες του σχεδίου έκθεσης, του σχεδίου μάλλον ψηφίσματος. Έχετε στο φακελό σας και το σχέδιο ψηφίσματος και τις τροπολογίες. 59 τροπολογίες είναι. Η συγητής μας, μόνιμος για το Βιετνάμ, είναι ο συνάδελφος Γιάν Ζαχράντιλ. Θα του δώσω λοιπόν το λόγο για να μας σχολιάσει τις τροπολογίες. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, με εν συντομία. Να σας επαναλάβω ότι εδώ έχουμε ένα σχέδιο ψηφίσματος για την ε, κατάσταση πρόοδου των ε, διαπραγματεύσεων για μια συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών με το Βιετνάμ. Ήδη έχουν ολοκληρωθεί έξι γύροι διαπραγμάτευσης. Θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαίωσε την πρόθεσή της να προβεί σε δήλωση για την πρόοδο των διαπραγματεύσεων αυτών στην ε, Σύνοδο Λομέλειας του Μαρτίου. Και βέβαια και η δική μας Επιτροπή πρέπει να εκφράσει την άποψή της να έχει λόγο για αυτό το θέμα. Μεταξύ άλλων γιατί είναι υποχρεωτική η έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για αυτή τη Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών. Αυτό σημαίνει ότι οι απόψεις μας είναι πολύ σημαντικές. Όπως προαναφέρατε κι εσείς, 59 συνολικά είναι οι τροπολογίες που κατέθεσαν οι συνάδελφοι, Σκιώδης και άλλοι. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για τη συμβολή τους και το πολύ επικοδομητικό πνεύμα που επέδειξα. Συν, ε, μάλλον διαπραγματευτήκαμε 10 συμβαστικές και 6 προφορικές τροπολογίες και μπορείτε να βρείτε τη σχετική διατύπωση και στον ε, τελικό κατάλογο ψηφοφορίας που έχει διανεμηθεί. Άρα το μόνο που μπορώ να κάνω τώρα εγώ είναι να ευχαριστήσω όλους όσους συμμετείχαν για τη θετική του στάση, για τη συμβολή τους και να παρακαλέσω τους συναδέλφους να στηρίξουν αυτό το σχέδιο ψηφίσματος για να μπορέσουμε να ψηφίσουμε στην Ολομέλεια του Μαρτίου. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Να ακούσουμε τους σκιώδες εισηγητές ή άλλα μέλη της Επιτροπής. Μπεντ Λάγκε. Ο σκιώδης από το ΕΛΚ είναι ο πρώτος που έχει το λόγο. Σοσιαλιστής. Τους σοσιαλιστές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ ιδιαίτερα και τον εισηγητή για την ε, σκεγράφηση των διαπραγματεύσεων, ιδίως για και για την εξαγωγή των διαπραγματεύσεων καθώ και ιδίω βέβαια για τις ε, τροπολογίες και τι συμβαστικές τροπολογίες. και την προσπάθεια να αναχαιτιστεί το παράνομο εμπόριο με εξωτικά είδη ζώων και φυτών. Νομίζω ότι η έκθεση που ψηφίσαμε τελικά είναι καλή. Δυστυχώς δεν υποστηρίζουν τις συμβαστικές τροπολογίες όλες οι πολιτικές ομάδες. Αυτό πιθανόν να οφείλεται και στο ότι επίκυνται οι ευρωεκλογέ. Ευχαριστώ πάντως ε, κύριε Πρόεδρε. Άλλος κανείς? Όχι. Ας ακούσουμε την Κομισιόν, αλλά φαίνεται πως η Κομισιόν δεν είναι ε, παρούσα, δεν έχει αποστείλει εκπρόσωπο. Συγητής, ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά όλους όσους ε, συμμετείχαν και κατέθεσαν τροπολογίες. Παναλαμβάνω ότι Είμαι και εγώ αισιόδοξο και όπω και ο κύριο Λάγκη ελπίζω αυτό το σχέδιο ψηφίσματο να τύχει θετική ψήφου αργότερα στην ψηφοφορία στην Επιτροπή. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος σας ευχαριστούμε. Θα ψηφίσουμε λοιπόν στην Ολομέλεια. Ελπίζουμε να επιβεβαιωθεί ότι θα γίνει αυτό τον Μάρτιο και περνάμε στο σημείο 13. Έχουμε λοιπόν την ώρα της ψηφοφορίας. Θα διακόψουμε μέχρι τις 10.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

Cristiana, benvenuta. Grazie. Ah, Cristina. Okay. buongiorno. Colleagues, welcome again. Good morning. Voting time. Συνάδελφοι, είναι η ώρα για τις ψηφοφορίες. Είστε έτοιμοι? Το πρώτο σημείο είναι το σημείο 13. Η μακροοικονομική συνδρομή στην Τινησία. Ας αρχίσουμε με την τροπολογία 6. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, τροπολογία 7. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 8. Υπέρ. Κατά αποχές έλεγχος. Ψηφίζουμε. Τέλος ψηφοφορίας. Τροπολογία 4 πρώτο τμήμα υπέρ, δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροποποιημένη λοιπόν η πρόταση της Κομισιόν ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Τέλος της ψηφοφορίας. Έγκρινεται με 20 ψήφους υπέρ και 3 κατά. Ε, τώρα ψηφίζουμε για το σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος ηλεκτρονικά. Τέλος της ψηφοφορίας. 21 ψηφί υπέρ, 2 κατά, καμία αποχή. Προτείνω να ξεκινήσει λοιπόν ο άτυπος ε, τριμερής διάλογος με το Συμβούλιο. Η εντολή έχει οθετηθεί και η σύσταση της διαπραγματευτικής ομάδας ως ήθιστε είναι, είμαι εγώ ως ε, ε, πρόεδρος και Συγητής, η κυρία ε, Σκάκελερ. objection? No, we need... Έχει κάνει αντίρρηση, όχι, ωραία. Ας ψηφίσουμε λοιπόν ηλεκτρονική ψηφοφορία. Τέλος της ψηφοφορίας. 21, μία ψήφι υπέρ, δύο αποχές, μία κατά. Εγκρίνεται. Επόμενο θέμα είναι το 14. Έχουμε έναρξη της ψηφοφορίας. Ο εισηγητής είναι Γιούλιο Βίνκλερ. Τέρας της ψηφοφορίας. 25 υπέρ, ένας κατά, Συγχαρτήρια. Και αυτό αφορούσε την συγκατάθεση για το πρωτόκολλο. Τώρα έχουμε κανονισμό για τη Σερβία. Σημείο 15 ψήφισμα για την κατάσταση προοδού για όσον αφορά τη Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών ΕΕ Βιετνάμ. Ο εισηγητής είναι ο κ. Ζαχαραντήλ, εξ ονόματος της ΙΝΤΑ. Υπήρχαν διάφορες τροπολογίες, αλλά ο εισηγητής μπόρεσε να τις ενσωματώσει σε συμβιβαστικές τροπολογίες. Να ψηφίσουμε λοιπόν τροπολογία 1 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. number Τροπολογία προ... Ε, προφορική 1 του εισηγητή, δεν υπάρχει αντίρρηση. Έχετε το προφορική νομίζω στο φάκελό σας. Ας ψηφίσουμε. Τροφορική τροπολογία του εισηγητή. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Υπέρ... Α, καταπίπτει. Παραμέντμαντ recital DA. Προφορική 2 στο αιτιολογική σκέψη DA. Υπάρχει αντίρρηση? Α, μάλιστα. Χρειάζομαι δύο που να έχουν αντίρρηση σύμφωνα με τον νέο, το νέο κανονισμό. Ένσταση. Που να έχουν ένσταση. One hundred fifty six in committee. 156 στην Επιτροπή είναι οι ψήφοι που χρειάζονται για να υπάρξει ένσταση κατά μιας ολομέλειας κτλ. κτλ. Άρθρο 156. Μα έχει ψηφιστεί στην Ολομέλεια, δεν έχετε κανένα δικαίωμα, όχι. Παρακαλώ. Η ένστασή σας λοιπόν δεν γίνεται αποδεκτή. Αυτό έχει ψηφιστεί στην Ολομέλεια και σας έχουν σταλεί. Ε, ε κοιτάξτε, οφείλετε να γνωρίζετε τους κανόνες και τους νόμους, ιδιαίτερα οι ευρωβουλευτές. Άρα λοιπόν η ένστασή σας δεν γίνεται αποδεκτή, απορρίπτεται. Λοιπόν, η προφορική, θα ψηφίσουμε την προφορική. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ελεκτρολικός έλεγχος για την προφορική τροπολογία. And vote is closed. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 15 υπέρ, 13 κατά. Καμία αποχή. Τροπολογία 4. Υπέρ, κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 6 Α, η 5, ναι, ναι, συγγνώμη. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 6, σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα ποιο είναι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 7, υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 10. Περνάμε στο, στην αντιλογική I. 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αν ελέγξουμε τη 10, μάλιστα, ηλεκτρονικός έλεγχος. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία στην αιτιολογική σκέψη J. Υπάρχει αντίρρηση σε αυτή την προφορική τροπολογία. Όχι. Ωραία. Ας ψηφίσουμε λοιπόν την προφορική ποιοι είναι υπέρ, κατά, εποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 13 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 14 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τροπολογία 17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 18 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται 19 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 26 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. να ελέγξουμε ηλεκτρονικά μάλιστα. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβαστική υπαριθμών 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην τροπολογία 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 34 είναι συμβατή. Ποιοι είναι υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Προφορική τροπολογία στην παράγραφο 9. Υπάρχουν αντιρρήσεις, ενστάσεις, όχι. Ε, ωραία, ας ψηφίσουμε λοιπόν. Προφορική 4, υπέρ κατά αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 37, υπέρ κατά αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 44 σε τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα, ποιοι είναι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα υπέρ, κατά αποχές... Α, έχει καταπέσει. Μάλιστα. Συμβιβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Προφορική υπαριθμών 5. Έχετε αντιρρήσεις? Όχι. Ας ψηφίσουμε. Ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Όχι, καλύπτεται από την προφορική 5. Κάποιοι θέλουν να το ψηφίσουμε. Ας ψηφίσουμε για τη 49, υπέρ, κατά, αποχές, Κοιτάξτε, αυτή ήταν η δική μου παρατήρηση ότι εφόσον καλύπτεται δεν χρειάζεται να ψηφίσουμε. Εγώ ακολουθώ τι μου λέει η γραμματεία. Ε, νομίζω ότι έχω δίκιο. Αν καλύπτεται, δεν χρειάζεται να το ψηφίσουμε. Λοιπόν, 51 έχουμε κατά τμήματα. Α, ναι, 50, σωστά. 50. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, Νομίζω πως ε, απερίφθη, αλλά ας, ελέγξουμε ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος της ψηφοφορίας. Απερίφθη. 51 κατά τμήματα ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Προφορική 6 υπάρχουν αντιρρήσεις. Ας ψηφίσουμε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 56. 56 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 57 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 58 οριστή ψηφοφορία πόσα τμήματα έχουμε 5 τμήματα Ωραία, ψηφίσουμε το πρώτο τμήμα. Της 58. Υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τρίτο τμήμα. γιατί το δεύτερο τμήμα έχει καταπέσει. Τρίτο τμήμα. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τέταρτο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 59 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Σχέδιο ψηφίσματος ε, όσο, όπως τοποποιήθηκε ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται λοιπόν με συντριπτική πλειοψηφία, 25 ψήφοι υπέρ, 2 κατά, 1 αποχή. Ε, συγχαρητήρια στον εισηγητή, τον κύριο Ζαχραντήλ. Σημείο 16. Έχουμε εδώ την ε, έγκριση των αποτελεσμάτων των διαπραγματεύσεων, των τριμερών διπλωματεύσεων με το Συμβούλιο και το Κομισιόν για τις, ε, τους διεθνείς εμπορικούς κανόνες. Ο εισηγητής είναι ο κ. Νινάλτη. Όσοι ήθιστε οι διαπραγματεύσεις μας βασίζονταν στην εντόλη, αλλά έπρεπε να γίνουν και συμβιβαστικές. Ε, οπότε τώρα χρειαζόμαστε τη δική σας έγκριση. μπορώ να σας πω ότι ήμουν παρόν και νομίζω πως πολύ καλά τα κατάφεραν ο εισηγητής μας. Εγώ συστήνω λοιπόν να εγκρίνουμε το αποτέλεσμα, ας ψηφίσουμε ηλεκτρονικά, τέλος της ψηφοφορίας. 28 υπέρ, ομοφωνία, καταπληκτικά τα καταφέρατε κύριε Ρινάλδη. Πολύ σημαντικός ε, ε, ο κανονισμός αυτός ώστε να αποκτήσει ε, κοφτερά δόντια η Ένωση. Περνάμε στο 17, έγκριση των πορισμάτων των τριμερών διαπραγματεύσεων. Πολ Μέρφυ, ο για την τροποποίηση του κανονισμού σε σχέση με τις αγωγέ ρυζιού καταγωγή Μπαγκλαντέ. Να ψηφίσουμε λοιπόν. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. 27 votes in favor. 27 Ψήφι υπέρ, καμία ψήφος κατά και μία αποχή. Συγχαρητήρια στον Πολ Μέρφυ. Ήμουν και εγώ εκεί. Item 17A. Um, uh, Πηγαίνουμε τώρα στο 17α. Όπως ξέρετε στην Ολομέλεια ψηφίσαμε τις τροπολογίες ε, στη πρόταση της Κομισιόν σε τέφα τον εξυγχρονισμό του CTI. Και θα πρέπει να ψηφίσουμε τώρα για την έναρξη των διαπραγματεύσεων του Συμβούλιο, να καθορίσουμε την εντολή, δηλαδή για αυτές τις τροπολογίες που εγκρίθηκαν στο Λομέλη και να αποφασίσουμε ποια θα είναι η σύνθεση της διαπραγματευτικής ομάδας που ως θα απαρτίζετε από τον πρόεδρο, από τον εισηγητή κύριο Φιέλνερ, Γιακολίνο, Σαρνέ, Στέρτη, Ζαντό, Σόλτς, Σαλβίνη. Ψηφίζουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. And what is... 25 ψήφοι υπέρ, καμία ψήφος κατά, μία αποχή. Και θα ξεκινήσει ο τριμερής διάλογος λοιπόν. Και εδώ ολοκληρώνεται η ώρα των ψηφοφοριών. Να ευχαριστώ όλους και όλες για την παρουσία σας. Όποιοι θέλουν να αποχωρήσουν, παρακαλώ ησύχως και γρήγορα. Okay. It's Antonio Parenti from the Commission. Το επόμενο θέμα είναι ανταλλαγή απόψεων για τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ιαπωνίας. Uh, Ξέρετε ότι ξεκίνησαν πέρυσι αυτές οι διαπραγματεύσεις ε, και η εντολή μας ε, έχει ήδη οριστεί με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Έχουμε και τη μόνιμη ομάδα παρακολούθησης ε, για την Ιαπωνία. Με πρόεδρο τον κύριο Καζάκ, ο οποίος είναι εδώ. Έχουμε καλέσει τους ε, ε, προσώπους των ενδιαφερομένων Ο ένας είναι από την ε, Ένωση Αυτοκινητομηχανίας. Έχουμε και τη φαρμακομηχανία που εκπροσωπείται με την κυρία Καρβέλιο συγκεκριμένα. Πού είναι οι φίλοι μας, εκεί μάλιστα, μπροστά μου. Ας δώσουμε το λόγο καταρχάς στον κύριο Πέσλα από την αυτοκινητομηχανία. Για 10 λεπτά έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, σα ευχαριστώ που μα δίνετε σήμερα τη δυνατότητα να σα εξηγήσουμε τη θέση μα για το πώ έχει η διαπραγμάτευση των συμφωνιών των εμπορικών. Επειδή ήταν στο Τόκιο ο κύριος Μίλιγκτον, θα ήταν καλό να του δώσω το λόγο να σας παρουσιάσει τα πράγματα. Βεβαίως, βεβαίως, παρακαλώ έχετε το λόγο. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε, κύριε και κύριοι. Λέγομαι Άντωνη Μίλιγκτον και είμαι εκπρόσωπος της ΑΣΕΑ στην ε, Ιαπωνία. Χαίρομαι πολύ που έχω τη δυνατότητα και σε μια πολύ επίκαιρη χρονική στιγμή να σας μιλήσω για την κατάσταση πρόοδου στις διαπραγματεύσεις ε, συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών με την Ιαπωνία και τις επιπτώσεις που θα έχει στην αυτοκινητομηχανία. Όπως θα γνωρίζετε, μετά από 12 μήνες διαπραγματεύσεων, τον Απρίλιο φέτος αναμένεται να γίνει μια εξέταση της πρόοδου της Ιαπωνίας στους πρώτους 12 μήνες για την εφαρμογή των δεσμεύσεων. Πριν ξεκινήσουν οι πραγματές είχε γίνει μια διερεύνηση και είχαν ε, οριστεί ε, τα προβλήματα που έπρεπε να αρθούν η δασμολογικοί φραγμή και θέλουμε να δούμε τι πρόοδο έχει επιτελέσει η Ιαπωνία ε, τους πρώτους αυτούς μήνες. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω όμως ότι αυτή η δημιουργική άσκηση ε, για το χάρτη ε, αυτοκινητομηχανίας και την άρση των μη δασμολογικών φραγμών δεν καλύπτει όλους τους μη δασμολογικούς φραγμούς και ελπίζουμε οι εν λόγω αυτοί φραγμοί να καλυφθούν στο επόμενο ε, γύρο διαπραγματεύσεων, να αποφασίσει βέβαια το Συμβούλιο. Τα μέλη θα συνεχιστούν αυτέ οι διαπραγματεύσει. Αυτή λοιπόν η άσκηση κάλυπτε έξι τομεί βασικά, με πρώτον την εναρμόνιση μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Ιαπωνία, τη ασφάλεια των αυτοκινήτων, βάσει των διεθνών ε, κανονισμών ε, του ΟΗΕ που έχουν συμφωνηθεί στη Γενέβη. Για τη δική μας ε, σκοπιά είναι πολύ σημαντικό αυτό το πρώτο βήμα προς την επίτευξη ενός μείζωνος στόχου των διαπραγματεύσεων, δηλαδή οποιοδήποτε όχημα που έχει έγκριση τύπου στην Ευρώπη με βάση τους κανόνες των ΗΠΑ να είναι αποδεκτό στην Ιαπωνία χωρίς οποιαδήποτε άλλη έγκριση τροποποίηση κτλ. Δεύτερος τομέας που καλύπτεται από αυτή την ερευνητική άσκηση είναι τα λεγόμενα αυτοκίνητα K, K-cars, τα πολύ ελαφρά οχήματα δηλαδή, που είναι ε, μια δημιουργία του ρυθμιστικού συστήματος της Ιαπωνίας. That if it looks like a car... 600 κυβικά μόνο είναι. Ε, αν το δείτε, θα είναι περίπου ίδιο με ένα οποιοδήποτε άλλο αυτοκίνητο, απλά έχει λίγο περισσότερο θόρυβο. Κάνει πολύ λίγο περισσότερο θόρυβο. Τρίτος τομέας. Γενικές εξαιρέσεις. Για συμβατικά airbag, και συμβατικούς αερόσακους και αερόσακοι που χρησιμοποιούν συμπιεσμένο υδρογόνο. Και αυτά ουσιαστικά γίνονται δυνάμει νομοθεσία που σχεδιαστεί για άλλου σκοπού. Αν θέλουμε να προωθήσουμε τη μεγαλύτερη ασφάλεια των αυτοκινήτων και εισαγωγή να προωθούν ε, τεχνολογία βελτιωμένη στην Ιαπωνία, θα πρέπει να έχουμε αυτή την εξαίρεση. Τρίτο τομέα, εναρμόνιση, παγκόσμια εναρμόνιση του κύκλου δοκιμών για την αποδοτικότητα των καυσίμων και, και τα καυσαέρια δεξάμενες ε, υψηλής πίεσης. that... Και σχεδιασμός των κινητών. Όταν Από τότε που ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις έχουμε δει να υπάρχει πρόοδος ε, σε άλλους τομείς περισσότεροι, σε άλλους λιγότεροι. Αλλά στην παρούσα φάση είναι δύσκολο να καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα. Πέμπτος γύρος διαπραγματεύσεων ε, θα έχει ολοκληρωθεί πριν την πρώτη αναθεώρηση. Είναι δύσκολο να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι έχει επιτευχθεί πλήρω ικανοποιητική πρόοδο σε όλου του τομεί αυτού. Μα ικανοποιεί πάρα πολύ η πρόοδο για του αερόσακου. Για να έχουμε μια γενική εξαίρεση, το πετύχαμε αυτό. Επίσης σημαντική ήταν και η πρόοδος σε ό,τι αφορά την έγκριση των κανονισμών ε, του ΙΑ από την Ιαπωνία, 11 τομείς παραμένουν στο σύστημα έγκρισης τύπου της Ιαπωνίας, που δεν δέχεται η Ιαπωνία ένα πιστοποιητικό ΟΗΕ που εκδίδεται στο πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης τύπου. Δεν ε, συμφωνεί με τις εθνικές απαιτήσεις της ε, Ιαπωνίας. Όμως τους τελευταίους 12 μήνες δεσμεύτηκε η Ιαπωνία, ευτυχώς, να εγκρίνει τέσσερις από τους εκκρεμείς ε, κανονισμούς του ΟΗΕ. Οι δύο, ε, για τους δύο επίκειται συμφωνία σε ό,τι αφορά τον αρουσμένο κύκλο δοκιμών και ελπίζουμε στο μέλλον αυτό να οδηγήσει σε έγκριση εκ μέρους της Ιαπωνίας των κανονισμών που εμπίπτουν στους τομείς αυτούς. Η πιο σημαντική εξαίρεση αφορά τρεις κανονισμούς, όπου η Ιαπωνία προτείνει στη Γενέβη ε, τροποποιήσεις ε, των εφιστάμενων κανονισμών για να ληφθούν υπόψη οι εθνικές απαιτήσεις της Ιαπωνίας. Εμείς δεχόμαστε ότι οι κανονισμοί του ΕΕ θα πρέπει να δεχθούν, να γίνουν αποδεκτοί λαμβάνοντας υπόψη και την τεχνική πρόοδο. Δεν πιστεύουμε όμως ότι είναι σωστό και σκόπιμο οι κανονισμοί του ΟΗΕ να σχεδιαστούν, είναι σχεδιασμένοι για να ε, λαμβάνουν υπόψη εθνικές απαιτήσεις της Ιαπωνίας. Μόνο εάν καταδειχθεί βέβαια ότι αυτό θα οδηγούσε σε μεγαλύτερη ξεκαθαρή αύξηση της ασφάλειας. Μέχρι στιγμή τα στοιχεία που έχουν δώσει στη Γενέβη οι Ιάπωνες δεν είναι αρκετά για να πείσουν τα άλλα συμβαλόμενα μέρη, που δεν είναι μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και άλλε χώρε. Όπω η Ρωσία, η Νότια Αφρική, ότι η πρόταση τη Ιαπωνία για τροποποίηση των κανονισμών αυτών είναι η δέουσα. Είναι ένα ακριβέ θέμα αυτό, ε, που θα γίνει αντικείμενο τεχνικών συζητήσεων στη Γενέβη. Σε ό,τι αφορά τα K-Cars, τα πολύ ελαφρά αυτά οχήματα, μέχρι στιγμής έχουμε κάποια πρόοδο. Η Ιαπωνική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι με την επιφύλαξη έγκριση του Κοινοβουλίου της Ιαπωνίας από 1η Απριλίου του τρέχοντος θα υπάρξουν κάποιες αλλαγές στη φορολόγηση των οχημάτων στην Ιαπωνία για να αρχίσει να κλείνει το χάσμα ε, σε ό,τι αφορά το επίπεδο της φορολόγησης αυτών των οχημάτων και κάποιων άλλων ε, πολύ μικρών οχημάτων, compact cars. Καλό είναι αυτό το πρώτο βήμα. Αλλά βέβαια πολλά απομένουν να γίνουν ακόμη μέχρι ότου κλείσει εντελώς το κενό αυτό και να μπορέσουν και τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά οχήματα να ανταγωνιστούν τα ιαπωνικά K-cars. Θα γνωρίζετε ίσως ε, ότι το 40% και παραπάνω ε, το, της αγοράς επιβατικών αυτοκινήτων της Ιαπωνίας καταλαμβάνεται από αυτά τα K-Cars. Το 40% δηλαδή της εγχώριας αγοράς της Ιαπωνίας είναι ε, κλειστή σε ξένο ανταγωνισμό γιατί κανένας ξένος κατασκευαστής πόσο μάλλον ε, από την Ευρώπη, δεν παράγει ε, αντίστοιχα οχήματα που να πληρούν στις προδιαγραφές αυτών των ιαπωνικών οχημάτων και cars. Θα έπρεπε να μπορέσουμε όμως να έχουμε και εμείς πρόσβαση σε, ε, μίσους τους όρους σε αυτό το μερίδιο της αγοράς. Πολλά λοιπόν ακόμη πρέπει να γίνουν. Είναι αφαρεντικό όμως κύριε Πρόεδρε το ότι σημειώθηκε κάποια πρόοδος. Η ΑΣΕΑ επιφυλάσσεται να κρίνει ε, μετά από τους 12 μήνες, δηλαδή κατά πόσον η πρόοδος αυτή μπορεί να θεωρηθεί πλήρως ικανοποιητική. Πάντως, εκτιμούμε τις προσπάθειες που καταβάλει η Κομισιόν για το θέμα των αερόσακων. Ο κύριος Ντεχούχτε ο ίδιος ε, ανέλαβε πρωτοβουλία για να πει στους Ιάπωνες να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους. Αυτά είχα να πω. Σας ευχαριστώ. Πρόεδρος. Δηλαδή είστε συγκρατημένο αισιόδοξο, αν κατάλαβα καλά. Ρεαλιστικά αισιόδοξο, ρεαλιστικά αισιόδοξο. Uh, uh, Σωστά δηλαδή ερμήνευσα, μάλιστα. Κυρία Τραβέλιο τώρα. Έχετε το λόγο. Της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Φαρμακο βιομηχανιών υποθέτουμε. Σας ευχαριστώ που μας δίνετε την ευκαιρία να εμφανιστούμε ενώπιον σας σήμερα για να σας εξηγήσουμε τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Φαρμακοβιομηχανίας σε σχέση με την FTA της, με την Ιαπωνία. Εμείς λεγόμαστε FPA, εκπροσωπούμε 1100 φαρμακοβιομηχανίες 33 εθνικές οργανώσεις, ε, ομοσπονδίες και ένα σύνολο 700.000 εργαζομένων και βεβαίως έμεσα ε, εξασφαλίζουμε απασχόληση σε άλλες ε, τρεις με τέσσερις φορές τον αριθμό αυτό. Σημαντικό λοιπόν. Και το πλεόνασμά μας είναι της τάξης των 54 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτό δηλαδή που εξασφαλίζουμε στις ευρωπαϊκές οικονομίες. Η Ιαπωνία είναι βέβαια σημαντικός παίκτη. Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη αγορά φαρμάκων στην, στον κόσμο, ε, της τάξης του 12%. Γι' αυτό η συμφωνία που βρίσκεται υπό επαναδιαπραγμάτευση είναι πάρα πολύ σημαντική. η FPA έχει και ιαπωνικές εταιρείε μεταξύ των μελών της και υπάρχουν και θηγατρικές στην Ιαπωνία. Στο Τόκιο έχουμε ήδη ιδρύσει την FPA Japan από το 2002 και εκεί εκπροσωπούνται 24 καινοτόμες ευρωπαϊκές βιομηχανίες στην Ιαπωνία. Έχουμε υποστηρίξει την συμφωνία διότι θεωρούμε ότι προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες. Ορισμένες από αυτές είναι ότι θα προσεγγίσουν οι αγορές μας, θα δώσουν όθηση επομένως στην ανάπτυξη και όφελος στους ασθενείς με τη διευκόλυνση των συνεργασιών και με δημιουργία νέων ευκαιριών για πρόσβαση στις αγορές και για τις ιαπωνικές και για τις ευρωπαϊκές εταιρείες. Μπορούμε να βοηθήσουμε να φέρουν σημαντική καινοτομία. Και βεβαίως να ενισχυθεί και η έρευνα. Η συμφωνία προσφέρει ακόμα την ευκαιρία να προχωρήσουμε σε ρυθμιστική σύγκληση, να καταργηθούν δηλαδή κάποιες προδιαγραφές οι οποίες αποτελούν εμπόδια για την ανάπτυξη. Έχουμε καλή συνεργασία με την Ιαπωνία σε πολυμερές επίπεδο υπό την αιγίδα της, διεθνής, της Διεθνούς ε, Συνόδου Εναρμόνισης Προδιαγραφών. Αυτό σημαίνει σημαντικό όφελος και για τους ασθενείς. Ωστόσο η FPA, η οργάνωσή μας, η μπορεί να αποτελέσει και την πλατφόρμα για την προώθηση ταχύτερης ρυθμιστικής εναρμόνισης. Στην συμφωνία θα θέλαμε να δούμε επέκταση της συμφωνίας για την αμοιβαία αναγνώριση των καλών παρασκευαστικών πρακτικών. Ήδη υπάρχουν οι σχετικές ρυθμίσεις και αυτές αναφέρονται σε όλα τα φαρμακευτικά προϊόντα και μεταξύ αυτών και στα εμβόλια. Αυτό είναι σημαντικό και για την προώθηση όλων των φαρμακευτικών προϊόντων στην Ιαπωνική αγορά. Και βεβαίως και να αρμοριθούν οι πολιτικές για τα εμβόλια για να καλυφθεί και το κενό εμβολίων που υπάρχει ακόμη και το οποίο δεν, ασφαλίζει, δεν εξασφαλίζει επαρκές, ε, επαρκές, επαρκές ποσότητες εμβολίων για τους ε, Ιάπωνες ασθενείς. Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οι ιδιαίτερες συνθήκες της αγοράς μας, να εξασφαλίζεται διαφάνεια και χώρος για καινοτομία η Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών τονίζει βέβαια και με ιδιαίτερο κεφάλαιο την ανάγκη προστασίας της διανοητικής ιδιοκτησίας και ότι τα μελλοντικά συστήματα θα ε, συμφωνούν, με, θα συμμορφώνονται με τις αρχές αυτές. Η, η βιομηχανία μας είπα ήδη ότι υποστηρίζει από την αρχή της διαπραγματεύσεις και θεωρούμε ότι πρέπει να ενισχυθούν οι προσπάθειες, διότι τα ενδεχόμενα ωφέλη από την Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών είναι σημαντικά. Κοινή δήλωση που υπογράφηκε στις 12 Νοεμβρίου του 2013 με την ευκαιρία της Ευρω-Ιαπωνικής Συνόδου Κορυφής 20 οργανώσεις, μεταξύ αυτών και η ΕΦΠΙΑ, επανέλαβαν την υποστήριξή τους για τη συνέχιση των συνομιλιών για να καταλήξουν σε μια συνολική συμφωνία. Αντιλαμβανόμαστε ότι οι διαπραγματεύσεις είναι περίπλοκες, δεν αποτελεί έκπληξη γι' αυτό για μας. Πιστεύουμε ωστόσο ότι έχει γίνει καλή προπαρασκευαστική εργασία εντοπισμού των ενωτήτων που πρέπει να αντιμετωπιστούν εξ αρχής. Και εμείς οι ίδιοι. Έχουμε αξιολογήσει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί ως τώρα. Εντοπίζουμε σημαντική πρόοδο σε ορισμένα από τα θέματα. Για παράδειγμα, για τις διατάξεις που έχουν σχέση με κλινικές δοκιμασίες για να φέρουν το ιαπωνικό σύστημα σε μια ευθυγράμμιση με τα συστήματα που προτείνει ο ICH και για άλλους τομείς βέβαια εκεί έχει υπάρξει λιγότερη πρόοδος για την MRA, για την κάλυψη του κενού των εμβολίων. Εκεί έχουν γίνει μικρά βήματα προς τη σωστή όμως κατεύθυνση. Και γι' αυτό εξακολουθεί να μας ενδιαφέρει η δυνατότητα να προχωρήσουν και ενθαρρύνουμε λοιπόν τους διαπραγματευτές να συνεχίσουν να επιδιώκουν τους στόχους αυτούς. Η πολιτική αξιολόγηση θα γίνει αργότερα φέτος, μετά από ένα έτος δηλαδή διαπραγματεύσεων. Και θα είναι σημαντική ευκαιρία να εξετάσουμε την πρόοδο που θα έχει επιτευχθεί ως τότε και να ενισχύσουμε και την πολιτική δέσμευση για την προώθηση μιας συνολικής και σε βάθος συμφωνίας για την ε, ελευθερία των συναλλαγών. Σας ευχαριστώ που μας επιτρέψατε να συμμετάσχουμε στην συνέδρια σας. Άρα λοιπόν τα βλέπετε θετικά τα πράγματα. Ναι, όντως και πιστεύουμε ότι θα γίνει καλή πρόοδος στις διαπραγματεύσεις. Σε ορισμένες από τις ενότητες έχει σημειωθεί αργή πρόοδος. Ωστόσο θεωρούμε ότι πρέπει και μπορούν να προχωρήσουν ταχύτερα. Σημειώστε τις ενδεχόμενες ερωτήσεις γιατί θα έχετε την ευκαιρία να απαντήσετε Μου σημειώνουν εδώ ότι ο κύριος Αντώνιο Παρέντη, αναπληρωτής επικεφαλής των διαπραγματεύσεων, είναι παρόν ως εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τώρα έχουμε τον Μετίν Καζάκ, που είναι επικεφαλής της ε, διαρκούς ομάδας παρακολούθησης. Μετίν, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, όπως ξέρετε, φτάνουμε στη στιγμή της ε, απογραφής των αποτελεσμάτων των διαπραγματεύσεων με την ταξί της Ένωσης και του της Ιαπωνίας. Πρέπει λοιπόν να δούμε μετά από πέντε γύρους διαπραγματεύσεων που έγιναν στις ριξέλες και στην Ιαπωνία Σήμερα στόχος μας είναι να ορίσουμε τη θέση του Κοινοβουλίου σε σχέση με αυτές τις εμπορικές διαπραγματεύσεις. Όπως ε, θα θυμάστε, στις 28 Οκτωβρίου 2012 το Ευρωκοινοβούλιο στήριξε την ε, ε, διαπραγματευτική εντολή γιατί είπαμε ότι ήταν σημαντικό να ενισχύσουμε τις σχέσεις μας με μεγάλους εμπορικούς εταίρους όπως η Ιαπωνία. Στόχος ήταν να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε την διερεύνηση με θετικό τρόπο και για τα δύο μέρη. Τα αποτελέσματα αποτελούσαν ένα βήμα μπροστά. Είπαμε επίσης ότι η εφαρμογή αυτής της δέσμευσης είναι πολύ σημαντική. Ε, θέλουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα ως προς αυτόν. Λοιπόν, όσο γινόταν πιο σύντομα. Επιπλέον το Κοινοβούλιο επέμεινε ότι η ε, ρήτρα αναθεώρηση θα έπρεπε να ενεργοποιηθεί ένα έτος μετά την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Ε, εμείς ζητήσαμε να, δοθούν, να, να υπάρχουν συγκεκριμένα αποτελέσματα όσον αφορά την κατάργηση μη, εμπορικό, μη τελωνιακών δασμών, ε, ιδιαίτερα όσον αφορά βασικούς τομείς της, ε, του εμπορίου όπως η οδικές αλλά και οι σιδηροδρομικέ μεταφορές οι οποίες συμπεριλήφθησαν στην ε, άσκηση διερεύνηση. Φτιάξαμε λοιπόν 21 οδικού χάρτες για τα μη δασμολογικά μέτρα ε, κατά τη γνώμη μου, η αξιολόγηση όλων αυτών των δικών χαρτών θα πρέπει να περιλαμβάνεται στην αναθεώρηση, καθώς καλύπτουν διάφορα θέματα στην αυτοκινητοβιομηχανία, στη χημική βιομηχανία, στην βιομηχανία τροφίμων, στη φαρμακοβιομηχανία, στις κατασκευαστικές εταιρείες, αλλά και ε, στους σιδηροδρόμους. Μιλήσαμε για αποτελεσματικούς ε, μηχανισμούς διευθέτησης ε, διαφορών, αναγνώριση γεωγραφικών ενδείξεων, ισχυρή και φιλόδοξη βιώσιμη ανάπτυξη και ένα σχετικό κεφάλαιο, καθώς και ένα κεφάλαιο για τις επενδύσεις. Δεν πιστεύω ωστόσο ότι θα πρέπει να δούμε μόνο τον καθρέφτη προς τα πίσω, αλλά να έχουμε μια γενική εξελόγηση της κατάστασης, γιατί όλες οι εξελίξεις που υπήρξαν θα πρέπει να ληφθούν υπόψη σοβαρά. Στις επόμενες εβδομάδες ε, σκοπεύω μαζί με τους συναδέλφους στην ε, ομάδα παρακολούθησης να συζητήσω με την Κομισιόν και τους ε, εμπλεκόμενους φορείς ώστε να μπορέσουμε να διατυπώσουμε τη θέση μας σε σχέση με την κατάσταση προόδου των διαπραγματεύσεων. Ε, λόγω του επικείμενου τέλους της θητείας μας, ε, στόχο έχουμε τα αποτελέσματα του προβληματισμού μας να κατατεθούν σε ένα ψήφισμα πριν το τέλος της θητείας μας. Είμαι ευτυχής λοιπόν που σήμερα έχουμε την ευκαιρία να ξεκινήσουμε τον προβληματισμό σε σχέση με αυτές τις βασικές διαπραγματεύσεις, ανταλλαγή απόψεων που στην οποία προέβημαν με τους βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς θα βελτιώσει την εργασία μας και πιστεύω ότι θα μπορέσουμε έτσι να αρχίσουμε να συζητάμε το θέμα από τις αρχές του Απριλίου. Ε, βέβαια η πρόοδος που έχει γίνει μέχρι τώρα είναι σχετικά περιορισμένη αλλά είμαι σχετικά ε, αισιόδοξο και ρελιστής και πιστεύω πως θα μπορέσουμε να δώσουμε στην Κομισιόν περισσότερα κίνητρα ώστε να πείσει την Ιαπωνική πλευρά να προβεί και να μάλλον σημειωθεί περισσότερη πρόοδο στον επόμενο γύρο. Η Κομισιόν δεν χρειάζεται κίνητρα, πρέπει απλά να τις πρόξουμε. Χρειάζεται όθηση. Όχι κίνητρα, τι να τους δώσουμε κίνητρα. Ας ακούσουμε τώρα τα υπόλοιπα μέλη της μόνιμης ε, Επιτροπής για την Ιαπωνία, τους αλλοσυγητές. Ο πρώτος είναι ο Γεροσλάφ Βαλένσα. Έλκα, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω μια ερώτηση προς την Κομισιόν. Τέσσερις μήνες πριν υπήρξαν κάποια θετικά σημάδια στις ε, συνομιλίες ε, για τις δημόσιες προμήθειες στον τομέα των σιδηροδρόμων. Το ερώτημά μου είναι, Πρόκειται για συστημική αλλαγή ή άπαξ έγινε, ε, υπήρξε αυτή η συμφωνία. Θα ήθελα κάποιες ε, διευκρινήσεις για τους διαγωνισμούς και το πώς ε, προχωρούν οι διαπραγματεύσεις με τις δημόσιες προμήθειες. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Επόμενος, ο υποφαινόμενος, γιατί είμαι σκιώδης για την ομάδα των σοσιαλδημοκρατών. Οπότε μιλώ υπό την ιδιότητά μου ως ε, μέλος ε, της ε, Επιτροπής και όχι πρόεδρος. Και εγώ πιστεύω ότι σημειώνουμε πρόοδο. Όμως μόνο η Κομισιόν έχει τη συνολική εικόνα. Πλησιάζει η ημερομηνία για την αναθεώρηση. δεσμεύσεις από πλευράς Ιαπωνίας ήταν πολλές. Πώς ε, κρίνει τα πράγματα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θεωρεί ότι εκπληρώνει τις δεσμεύσεις της η Ιαπωνία. Θα είναι θετική η αξιολόγηση. Θα το δούμε. Δεύτερον, θεωρούνται ευαίσθητα ορισμένα διατροφικά προϊόντα λόγω τη ε, ιαπωνικής ε, δίαιτα. Υπάρχουν κάποιες κόκκινες γραμμές ό,τι αφορά το άνοιγμα λοιπόν ε, το εμπορικό και το βόλιο κρέα, το χείριο κρέα, τα γαλακτοκομικά προϊόντα, το ρύζι, το στάρι, το άμυλο, ε, η ζάχαρη και το κρυθάρι είναι μεταξύ αυτών των προϊόντων. Η Κομισιόν πώς ε, εκτιμά την κατάσταση. Θα μπορούσε αυτό να περάσει αρνητικά τις διαπραγματεύσεις σε αυτή τη φάση. Θα μπορούσε ίσως να αλλάξει κάτι στο μέλλον. Νομίζω πρέπει να λάβουμε μια απάντηση στο ερώτημα αυτό. Τώρα, ευρύτερα, για τη συμμετοχή της Ιαπωνίας στις διαπραγματεύσεις ε, TPP. Αποφάσισαν να προσχωρήσουν ε, σε ε, ύστερο στάδιο της διαδικασίας διαπραγματεύσεων που έχουμε με του ΣΥΠΑ και τους άλλους μας εταίρους από τον Ειρηνικό. Η προσχώρηση λοιπόν της Ιαπωνίας στο TPP τι επιπτώσεις θα μπορούσε να είχε. θα μπορούσαν να περαστούν οι δεσμεύσεις τους να είναι σε διαπραγματεύσεις μαζί μας, εάν δηλαδή υποχρεωθούν να κάνουν επιλογές, να επιλέξουν κάτι. Τι θα επιλέξουν. They are also negotiating... Uh, Τέλος, είναι και ανοιχτή στο ενδεχόμενο διαπραγμάτευση τριμερού συμφωνίας με Κίνα και Νότια Κορέα. Τι αντίκτυπο θα μπορούσε να έχει αυτό. Ήδη έχουν πολύ στενές εμπορικές σχέσεις αυτές οι τρεις χώρες και βέβαια αυτή η συμφωνία θα εμβαθύνει και θα διευρύνει την ε, ολοκλήρωση των τριών αυτών οικονομιών. Τι επιπτώσεις θα μπορούσε να έχει αυτό. για το δυναμικό των δικών μου μας ε, συμφωνιών. Χρειαζόμαστε, πιστεύω, μια πιο συνολική εικόνα και η Κομισιόν φαντάζομαι ότι έχει τα στοιχεία και τις πληροφορίες για να μας ε, μεταφέρει. Επόμενος ε, σκιώδης. Ποιος είναι? Από την ομάδα ECR δεν βλέπω το σκιώδη. Next one is Helmut. Άρα, ο από την ΚΟΥ, ο κύριος Helmut Σόλτ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ επίσης Ευχαριστώ επίσης και τους εκπροσώπους των βιομηχανιών που εξήγησαν την δική τους σκοπιά. Αλλά έχω και τρία κάπως ευρύτερα σχόλια για τις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις. Θα ήθελα επίσης να ακούσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το πού βρισκόμαστε στον τομέα των προμηθειών, δημοσίων προμηθειών. Η υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί στην πρόοδο που έχει γίνει. Πού βρίσκεται λοιπόν η κατάσταση στον τομέα των δημόσιων προμηθειών. Το ίδιο με τις υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες του χρηματοπιστωτικού τομέα ο έλεγχος του χρηματοπιστικού τομέα που είναι σημαντικός και για τις δύο πλευρές. που είναι σημαντικός και για το ξεπέρασμα της κρίσεως και στην Ευρώπη και στην Ιαπωνία βέβαια. Συχνά ακούγονται σχόλια περί ρυθμιστικού πλαισίου Τι μπορεί να μας πούν για αυτό το τομέα της συμφωνίας. Το ίδιο με ενδιαφέρει ο προβληματισμός για την TPP και ιδίως μετά από την ανακοίνωση των Ιαπώνων ότι αρχίζουν να συμμετέχουν στην διαδικασία TPP επειδή όμως τότε σημειώνονται ευρύτερα προβλήματα για την TPP, αυτή έχει αρχίσει και επιβραδύνει. Τι γίνεται επίσης για τις σχέσεις μεταξύ Ιαπωνίας και Κίνας, διότι και η Κίνα ενδιαφέρεται να έχει πρόσβαση στις διαπραγματεύσεις TPP. Και έρχομαι στο τρίτο ερώτημα. Προχωρούμε τώρα στις διαπραγματεύσεις για τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Κίνας και τις επενδύσεις. Το κεφάλαιο των επενδύσεων για, με τους Ιάπωνες δηλαδή, τι ρόλο θα παίξει και το ίδιο ο μηχανισμός διευθετήσεως διαφορών. Ευχαριστώ αγαπητέ Σόλτς. Εσείς τώρα έχετε το λόγο, χωρίς μικρόφωνο. Έχω λεπτομερείς ερωτήσεις. Και αν δεν γνωρίζετε τις απαντήσεις, να μου τις στείλετε γραπτός. Υπάρχει ήδη συμφωνία μεταξύ Ελβετίας και Ιαπωνίας. Ερώτηση. Ποιες είναι οι ρήτρες εκείνες στην συμφωνία Ελβετίας-Ιαπωνίας που θα είναι ενδεχόμενα απαράδεκτες για τους Ευρωπαίους διαπραγματευτές. Δεύτερη ερώτηση για το ίδιο θέμα. Ποιε ρήτρε στην ίδια συμφωνία Ελβετίας Ιαπωνίας. Επιθυμούν ενδεχομένω οι Ευρωπαίοι διαπραγματευτές να βελτιώσουν. Αν δεν γνωρίζετε τις απαντήσει ήδη τώρα μπορείτε να μου τις αποστείλετε γραπτός. Μα με την, με την ε, Ελβετία συναγωνιζόμαστε τώρα. Λέει ο Πρόεδρος. Η Ελβετία είναι το όροσημό μας, το benchmark. Νομίζω ότι κάπως τελευταία έχουν αποδείξει ότι δεν είναι. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πολλά θέματα σας έθεσαν υπόψη. Κύριε Παρέντη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είμαι πολύ ευχαριστημένος με τους θετικούς απόϊχους που είχα από τους ενδιαφερόμενους φορείς αλλά και από τον εισηγητή τον κύριο Καζάκ. Πιστεύω πως σαφώς επέδειξε τα προσπάθεια που κατέβαλε η Κομισιόν για να συνεργαστεί στενά με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς και για την ε, συνελλογή πληροφοριών και την καταγραφή ε, ιεράρχηση προτεραιοτήτων. Ε, έγινε πολύ πρόοδος λοιπόν αυτή την πρώτη ε, χρονιά. Σίγουρα είναι εντυπωσιακή σε σχέση με το ποια ήταν η κατάσταση των σχέσεών μας ε, ε, όσον αφορά πούμε, τα διάφορα μέτρα πριν ξεκινήσουμε αυτές τις ε, διαπραγματεύσεις. Τώρα σημαίνει αυτό ότι είμαστε στο τέλος των διαπραγματεύσεων. Όχι βέβαια. Αυτό που σημαίνει είναι ότι βλέπουμε θετικά αυτές τις πρώτες ε, διαπραγματεύσεις και την πρώτη αυτή συντονισμένη προσπάθεια για ε, να λάβει, για να ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις που ανέλαβε η Ιαπωνία στην πρώτη προσπάθεια διερεύνησης των ε, στόχων μας. Βεβαίως, και θα συνεχίσουμε να ζητούμε την επίτευξη αυτών των στόχων αν μπούμε σε δεύτερο γύρο ε, διαπραγματεύσεων. Θα πρέπει να διαπιστώσουμε ότι και να καταγράψουμε ότι έγιναν πολλές προσπάθειες στη συζήτηση αυτών των θεμάτων μέχρι στιγμής και νομίζω ότι ε, έγιναν και παρατηρήσεις ε, για τη τελευταία τελική μάλλον συμφωνία όπου έχουμε προβλήματα. Υπάρχουν διάφορα κεφάλαια όπου πρέπει ακόμα να γίνει αρκετή δουλειά μετά από τέσσερις γύρους ε, διαπραγματεύσεων. Και αυτά θα τονιστούν περισσότερο στο μέλλον, ε, ας πούμε βιώσιμη ανάπτυξη. Είναι ανάμεσα στα θέματα που θέλουμε να τονίσουμε περισσότερο και να έχουμε πιο θετικά αποτελέσματα στη συνέχεια. Η αναθεώρηση που θα γίνει μετά από τον πέμπτο γύρο θα αρχίσει τον Απρίλιο ε, στο Τόκιο και σίγουρα, όπως είπε και ο κύριος Καζάκ, θα απαιτήσει μια σαφή αποτίμηση της κατάστασης για την εφαρμογή των συμφωνιών ε, αλλά και μια γενική αξιολόγηση για το πού βρίσκεται η κατάσταση των θα εξετάσουμε όλα τα στοιχεία, ιδιαίτερα το στοιχείο της πρόσβασης στην αγορά που θα εξακολουθήσει να είναι σημαντικό για μια χώρα όπως η Ιαπωνία που έχει χαμηλότερες δασμούς για πολλά προϊόντα αλλά και ψηλότερους δασμούς για πολλά από τα προϊόντα της ευρωπαϊκής επιθετικής ε, βιομηχανίας. Συνεργαζόμαστε με το Κοινοβούλιο και τον κύριο Καζάκη να διευκολύνουμε τον το σχηματισμό θέσης από πλευράς του Κοινοβουλίου. Τώρα, σε σχέση με την συμμετοχή των Ευρωβουλευτών, υπάρχουν θέματα για τις δημόσιες συμβάσεις. Εδώ νομίζω δεν σας πω καλύψω κανένα μυστικό. Αν σας πω ότι είναι ένα από τα πιο περίπλοκα θέματα που διαπραγματευόμαστε με την Ιαπωνία. Ε, έχουν γίνει και εδώ κινήσεις. Είναι περίπλοκη η διαπραγμάτευση λόγω της δομής της αγοράς των δημοσίων συμβάσεων, όπου η Ιαπωνία έχει τρεις βασικά μονοπολιστικές ιδιωτικές εταιρείες που αναλαμβάνουν όλα τα, τις δημόσιες συμβάσεις, αλλά είδαμε πως καταβάλλονται ισχυρές προσπάθειες από τους Ιάπωνες να προσπαθήσουν να εντοπίσουν να επιβάλλουν διαφάνεια στη λειτουργία της ρήτρα της επιχειρησιακής ασφάλειας που χρησιμοποιήθηκε στο παρελθόν για να εξαλειφθεί η δυνατότητα ανοιχτών ε, διαγωνισμών και η δυνατότητα ε, εφαρμογής των κανόνων ε, για αυτές τις εταιρείες. Θα πρέπει να δουλέψουμε πολύ μέχρι το τέλος της ετήσιας περίοδου αναθεώρησης. Τώρα, για τα γεωργικά προϊόντα, τα ευαίσθητα τα οποία εσείς ε, αναφέρατε, σε αυτούς τα προϊόντα αυτά είναι ε, σημαντικά για την Ένωση, όχι όλα, γιατί δεν είμαστε, ας πούμε, εξαγωγής ρυζιού αλλά σίγουρα είμαστε εξαγωγή ε, βοήου και χειρίου κρέατο. και αυτό το θέμα θα πρέπει να συζητηθεί με την Ιαπωνία γιατί αυτή τη στιγμή δεν συζητείται. Προσπαθούμε να καταλάβουμε ποια ακριβώ είναι η ευαισθησία τη Ιαπωνία σε κάποια θέματα, αλλά ευαισθησία σημαίνει και κάποιο βαθμό ευελιξία από πλευρά σου για να βρεθεί μια λύση που να είναι κατάλληλη και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω και αυτό δεν σημαίνει ότι θέλουμε να ε, τα αποφύγουμε στην ε, TPP, στην ε, διατλαντική εταιρική σχέση. Όχι. Υπάρχουν δυνατότητες εξαγωγών. Η Ιαπωνία θα οφείλει να βρει μια λύση για αυτά τα προϊόντα και σε αυτό το πλαίσιο. Και έτσι έρχομαι στο θέμα της συμμετοχής του TPP, ποιες, είναι, θα είναι οι πιθανές επιπτώσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εν γέννη, θεωρούμε πως οι δύο διαπραγματεύσεις είναι συμπληρωματικές σε κάποιο βαθμό έχουμε κοινέ απόψεις και στόχους. Υπάρχουν τομείς φυσικά όπου θα μπορούσαμε να καταλήξουμε σε προβλήματα δεν έχουμε απαραίτητα την ίδια δομή υποδομών όπως η ΕΠΑ, η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία για να αναφέρω απλώς κάποια από τα μέλη του, της συμφωνίας TPP της, ε, της ε, συμφωνίας με τις χώρες του Ειρηνικού αλλά κατά μέσο όρο ο Μόνο στο μέσο που υπάρχει κίνδυνος είναι ο τομέας των γεωγραφικών ενδείξεων, γιατί εμείς έχουμε διαφορετική ιδεολογία για αυτό το θέμα ανάμεσα στην Ευρώπη και τα περισσότερα μέλη της ε, συμφωνίας αυτής. Οι Ιαπωνές το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά αυτό. Νομίζω πως υπάρχουν πολλοί Ιάπωνες φορείς που εξετάζουν το ευρωπαϊκό σύστημα από μεγάλο ενδιαφέρον, ιδιαίτερα εφόσον θέλουν να απελευθερώσουν το γεωργικό του τομέα και αναμένεται ε, νέα νομοθεσία για τις ε, γεωγραφικές ενδείξεις και έχουμε συνεργαστεί μάλιστα με τους Ιάπωνες για να διευκολύνουμε τη σύνταξη, την κατάρτιση σχετικής νομοθεσίας που θα, μας, θα επιτρέψει βέβαια να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις μαζί μας αλλά και με τη, στο πλαίσιο της TPP. Τώρα, για τη συμφωνία που αναφέρατε με την Κίνα και την Κορέα. Το πρώτο που θα πρέπει κανείς να διερωτηθεί και που ειλικρινώς δεν έχω απάντηση είναι πόσο εις βάθος θα προχωρήσουν αυτές οι διαπραγματεύσεις, τι θα καλυφθεί πέρα από την απελευθέρωση του εμπορίου στα αγαθά και σε ποιο βαθμό, μέχρι πού θα προχωρήσουμε. Δεν είμαι βέβαιος ότι αυτή η συμφωνία θα έχει το ίδιο επίπεδο ε, φιλοδοξίες με αυτήν που διαπραγματευόμαστε μέσω του TPP. Σίγουρα όμως θα οδηγήσει σε περισσότερη ολοκλήρωση στον τομέα. Κάποιες μέρες ε, πριν έγινε μία δήλωση από την BASF, νομίζω, την Ευρωπαϊκή Εταιρεία BASF, που σε ενδιαφέρον για εγκατάσταση ενός ερευνητικού κέντρου στην Ιαπωνία για να καλύπτει την ε, περιφέρεια Ασίας Σιρηνικού. Ε, η συμφωνία μας με την Ιαπωνία μαζί με συμφωνίες όπως αυτή που διαπραγματευόμαστε στο, στην περιοχή του ΑΣΕΑΝ θα διευκολύνει και τις δυνατότητες των εταιριών μας να ανταποκριθούν στις προσδοκίες μιας ε, οικονομικά αναπτυσσόμενης ε, Ασίας. Το θέμα τώρα της ρυθμιστικής συνεργασίας που μας ρωτήσατε για το θέμα το χρηματοπιστωτικό δεν είναι εύκολο καθόλου. Θα χρειαστεί περαιτέρω εξέταση από την πλευρά των Ιαπώνων και αυτό θα συμβεί μόνο εάν ε, δοθεί η διαπραγμάτευση. Υπάρχει τώρα κανένας αντίκτυπος στις σχέσεις μας με την Κίνα λόγω της επιβράδυνσης του TPP. Μακάρι να έχω να σας πω μια σαφή απάντηση. Πάντως υπάρχει πιθανότητα η Κίνα να κερδίσει κάποιο χρόνο και να προσπαθήσει ίσως να χρησιμοποιήσει το σύστημα μεταρρυθμίσεων που έχει αρχίσει για, ή να το επιταχύνει για να καταφέρει να ενισχύσει περισσότερο τις διμερείς σχέσεις με τις διάφορες χώρες, αλλά δεν βλέπω να υπάρχει μέγας αντίκτυπος σε αυτή την επιβράδυνση. Ούτε στη σχέση μας με την Κίνα, ούτε με την Ιαπωνία. Η Ιαπωνία ίσως να ενδιαφερθεί να προχωρήσει περισσότερο μαζί μας γιατί η πτυχή του TPP μπορεί να χρειαστεί να καθυστερήσει τουλάχιστον μέχρι τις αμερικανικές εκλογές. Τώρα, επενδυτική συμφωνία είναι τμήμα ε, των εμπροματευσεών μας. Εμείς ε, εξετάζουμε τις δυνατότητες ε, ανταλλαγής μια ε, προσφορά επενδύσεων κοντά στο πέμπτο γύρο, η συζήτηση για έναν μηχανισμό ρύθμισης των διαφορών ε, στο επενδυτικό κεφάλαιο βρίσκεται ακόμα στην αρχή. Ε, για την ώρα δηλαδή εξετάζουμε τις διάφορες επιλογές συμπεριλαμβανόμενε αυτής για το σύστημα επίλυσης διαφορών του κράτους επενδυτή. για την ε, συμφωνία Ελβετίας-Ιαπωνίας. Ειλικρινά δεν ξέρω τι είναι αποδεκτό και τι όχι. Εμείς ε, δεν χρησιμοποιήσαμε ως ορόσημο την συμφωνία με την Ελβετία. Με την Ελβετία η συμφωνία όσο και αν είναι σημαντική είναι σχετικά περιορισμένη σε σχέση με αυτό που θέλουμε να διαπραγματευτούμε. Δεν καλύπτει αρκετούς τομείς ε, πολύ μεγάλου ενδιαφέροντος για μας, ιδιαίτερα στο μη δασμολογικό τομέα και στις υπηρεσίες. Οπότε σκοπεύουμε να προχωρήσουμε περισσότερο. Ειλικρινά δεν έχουμε πάει άρθρο-άρθρο τώρα για να δούμε τι μπορούμε να ε, αντιγράψουμε όσο έχει και τι όχι. Θα πρέπει να προσαρμόσουμε εξάλλου την εντολή μα για να διαπραγματευτούμε την Ιαπωνία που είναι μια από τι σπουδαιότερε και μεγαλύτερε οικονομίε. Ελπίζω να απάντησα στι ερωτήσει. Σας ευχαριστώ. Να κλείσουμε. Και επανέρχομαι στους προσκεκλημένους μας αν έχουν να κάνουν κάποιο τελικό σχόλιο. Κύριε Μπέρζελεν. Um, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να πω λίγα λόγια. Ότι δηλαδή μια τέτοια συμφωνία ελευθερών συναλλαγών είναι μακροπρόθεσμη δέσμευση μετά από ένα χρόνο όντω τα πράγματα είναι σχετικά ρόδινα. Σύμφωνοι. Πρέπει να δούμε όμω ποιε θα είναι οι επιπτώσει τη FTA για διαφόρου λόγου. Εγώ δεν μπορώ παρά να συγκρίνω με τι εμπειρίε που έχουμε σήμερα από τη συμφωνία με την Νότια Κορέα. Η δική μου σύσταση προ του διαπραγματευτέ θα ήταν να πω κάνατε ό,τι μπορέσατε για να βάλετε ένα παράδειγμα για τα αυτοκίνητα που να έχει κάποιο νόημα. Σήμερα είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση διότι έχουμε υπαρκτά μη δασμολογικά εμπόδια τα οποία εξακολουθούν να ισχύουν. Πάτε στην Ιαπωνία τώρα να κάνει το ίδιο ο το και η δική μου σύσταση είναι να κάνετε κάθε δυνατή προσπάθεια για να υπάρξει μια κατάσταση όπου να μην χρειάζεται να ε, ασχολούμεθα καθημερινά με τρόπους για να λύσουμε τα προβλήματα που έχουμε με την Κορέα. Αυξάνουν οι εξαγωγές μας προς την Κορέα σημαντικά, λέει ο πρόεδρος. Απάντηση χωρίς μικρόφωνο. Υπάρχει μια αύξουσα δημοτικότητα των οικονομικών σε καύσιμα αυτοκινήτων. Έχουμε είναι τεράστια η αύξηση. Από 20.000 αυτοκίνητα πριν από λίγα χρόνια έχουμε φτάσει στα 80.000 αυτοκίνητα. Αλλά αυτό έγινε και πριν ακόμα συναυθεί η FTA. Ναι, αλλά ε, κοιτάξτε πώς πήγε η καμπύλη. Πάρα πολύ απότομα ανεβαίνει. Ναι, ωραία είναι αυτά, λέει ο πρόσωπος της Άσεα. δεν ξέρω βέβαια για πόσο καιρό θα συνεχιστεί. Μπαίνει όμως και ένα θέμα όπου μακροπρόθεσμα έχουμε ένα automotive annex, ένα παράρτημα για τα αυτοκίνητα δηλαδή, με παραθυράκια και που επιτρέπει την διατήρηση μη δασμολογικών φραγμών, καθώς και την προσθήκη νέων. Αντιλαμβάνομαι ότι ιδίω οι Γερμανοί τα πάνε πολύ καλά στην Νότια Κορέα σήμερα και ελπίζω αυτό να συνεχιστεί, αλλά οι μη δασμολογικοί φραγμοί υπάρχουν και όλοι οι υπόλοιποι θίγονται. μη δασμολογική φραγμοί, οι οποίοι μάλιστα προστίθεται νέοι και θα σας στείλουμε και λίστα άμα θέλετε. Βέβαια τίποτα δεν είναι τέλειο λέει ο πρόεδρος, η κυρία Τρεμπέλιο των φαρμάκων. Από τη δική μας πλευρά είμαστε πανέτοιμες να συνεργαστούμε με τον κύριο Καζάκ για την ε, εργασία της ε, Monitoring Group και θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που μας ε, προσέφερε μια επισκόπηση της προόδου που έχει επιτευχθεί ως τώρα καθώς και των προκλήσεων που μας περιμένουν στο μέλλον. Και να επαναλαμβάνω την υποστήριξή μας και πάλι και εμείς θα προσπαθήσουμε να συμβάλλουμε με τον τρόπο μας στην ε, πρόοδο των διαπραγματεύσεων. Ο κύριος Καζάκ ως μόνιμος εισηγητής. Ευχαριστώ για την ανταλλαγή απόψεων που δείχνει ότι όλοι ενδιαφερόμαστε να ειδούμε μια πραγματική πρόοδο στο ευαίσθητο αυτό θέμα. Με τους Ιάπωνες και επιθυμούμε να σημειωθεί μεγαλύτερη πρόοδος. Είναι βέβαια σαφές ότι δεν μπορούμε να επιτύχουμε όλα τα αποθούμενα, αλλά τουλάχιστον να έχουμε ικανοποιητικά αποτελέσματα. Και όλες οι δυνατότητες που έχει στη διάθεσή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να πείσει τους Ιάπωνες να προχωρήσουν σε μεγαλύτερη πρόοδο πριν από τον πέμπτο γύρο των ε, διαπραγματεύσεων. Όλα αυτά λοιπόν τα εκτιμώ. Αναμένω τη συνεργασία, ως συνήθως των εταίρων μας, των ενδιαφερομένων, των stakeholder δηλαδή, που συμμετέχουν στην ε, ομάδα παρακολούθησης και να γνωρίζουν βεβαίως, ε, να είναι ενήμεροι για την πρόοδο πριν από την ε, ολοκλήρωση της παρούσας θητείας. Μάλιστα, το επόμενο, το επόμενη φάση θα είναι συνάντηση με τον ίδιο τον Επίτροπο Ντεγκούχτ τον Απρίλιο. Το μήνυμά μας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι φανείτε σκληροί απέναντί τους και φέρτε μας μια καλή συμφωνία. Θέμα 19. Πρόοδος των ανεξελίξης τριμερών διαπραγματεύσεων. κανείς από τους εισηγητές, άρα θα μιλήσω εγώ. Αφού είχα πάει σε όλους άλλωστε τους τεμένους διαλόγους. Για τον κανονισμό χρηματοοικονομικής ευθύνης, ISDS, Πάβελ Ζαλεύσκη εισηγητής. Ε, ξέρετε ότι είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της νέας επενδυτικής πολιτικής της Ένωσης, όμως δεν έχω να σας δώσω δυστυχώς καλά νέα. Μήπως θα μπορούσα να ζητήσω από τους προσκεκλημένους μας να συνεχίσουν τις συνομιλίες τους εκτός της αίθουσας, παρακαλώ. Pictures of cards outside, please και η αλλαγή καρτών ε, επισκεπτηρίων λοιπά να γίνει εκτός της αίθουσας παρακαλώ. Για το ISDS λοιπόν, επαναλαμβάνω την ε, επίλυση διαφορών επενδυτή κράτους. Ε, δεν έχω να σας δώσω καλά νέα. Υπάρχει διαίρεση μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. Το χάσμα δεν έχει μειωθεί. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε ένα, ένα ανεπίσημο έγγραφο, ένα non-paper, το Συμβούλιο δεν συμφωνεί με αυτό το έγγραφο, εμείς θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε και άρα δεν υπάρχει εντολή σε επίπεδο Συμβουλίου. Άρα κρίμα, αλλά δεν θα μπορέσουμε μέχρι το τέλος της κοινοβουλευτικής περίοδου να έχουμε ολοκληρώσει. Γιατί για να έχουμε και μια ισχυρή επενδυτική πολιτική πρέπει να μπορούμε να πούμε στους εταίρους με τους οποίους δεν πραγματευόμαστε ότι θα γνωρίζουμε τελικά ποιος είναι υπεύθυνο υπόλογος για οποιαδήποτε ζημία. Και οφειλόμενοι από ζημιωσή όμως το Συμβούλιο δεν συμμερίζεται την ανησυχία μας. Είναι λοιπόν κάπως ανησυχητικά τα πράγματα και ιδίως ως προς το ότι το Κοινοβούλιο και η Κομισιόν ε, έχουν απόψεις που δεν συμμερίζεται το Συμβούλιο. Και μιλάμε εδώ για τις αρμοδιότητες κρατών μελών και ένωσης για την επενδυτική πολιτική. Η συνήθεια της Λισαβόνας δηλαδή ερμηνεύεται διαφορετικά από τους μεν και τους δε. Οπότε φαντάζομαι ότι η τελική λύση είναι να αποφασίσει το δικαστήριο για αυτή τη διαφορά. Ο τελικός κανονισμός εγκρίθηκε μετά από διαπραγματεύσει με το Συμβούλιο, με πολύ βοήθηση και συμμετοχή της Κομισιόν. Σημαντικός κανονισμός, γιατί έπρεπε να αναλαμβάνουμε ad hoc πρωτοβουλίες για να επιβάλλουμε μέτρα σε περίπτωση παραβιάζουν των εμπορικών δικαιωμάτων στο πλαίσιο των κανόνων του ΠΟΕ. αυτό είναι μια καλή είδηση. Εισαγωγή, δασμοί, αποπαντετές. ναι, πράγματι ήταν περιορισμένο το πεδίο, ολοκληρώσαμε, ήταν ένα κανονισμός ευθυγράμμισης ουσιαστικά. δική μας πρωτοβουλία εγκρίναμε και κάποιες τροπολογίες επί της ουσίας του κανονισμού. Ένας αποδεικτός εμπιβασμός εξευρέθη τελικά. Ένα άλλο θέμα. Διαχωριστική γραμμή μεταξύ εκταλιστικών και κατεξοδότηση πράξεων δεν το έχουμε ακόμη τακτοποιήσει το θέμα. Δεν έχουμε βρει ένα σαφή ξεκάθαρο ορισμό φιλοσοφία. Έχουμε την για πολύ καλή δουλειά. Βίβλος θα πρέπει να είναι για μας σε ό,τι αφορά τις εκτελεστικές και κατεξοδότητες πράξεις. Δεν φαίνεται όμως ε, όλοι οι συνάδελφοι από όλες τις άλλες επιτροπές να έχουν αντιληφθεί τη σημασία που έχει να υπάρχουν σαφή κριτήρια. Και βέβαια το Συμβούλιο το εκμεταλλεύεται. και πιέζει τα πράγματα προς φυσικά προς το συμφέρον του, προτιμά δηλαδή τις ε, εκτελεστικές από τις κατεξουσιοδότηση πράξεις. Δηλαδή προτιμά τη διαδικασία εξέτασης και όχι τη συμβουλευτική διαδικασία, τη γνωμοδοτική διαδικασία. Γίνεται πραγματική μάχη. Το Συμβούλιο φαίνεται αποφασισμένο να προσπαθήσει να ανακτήσει Κάποιε από τι αρμοδιότητες που έχασαμε με τη συνθήκη τη Λισαβόνα. Επικίνδυνη στάση. Και το Κοινοβούλιο δεν μπορούμε συστηματικά να χάνουμε αυτέ τι μάχε με το Συμβούλιο. σε ένα άλλο θέμα είχαμε θετική εξέλιξη, πάλι καθεξοδότηση πράξη ε, implementing ε, εκτελεστικές, no opinion clause, ε, ε, ρήτρα μη γνωμοδότηση κτλ. Αλλά νομίζω ότι είναι ένας ισορροπημένος συμβιβασμός με κάποιες απώλειες που δεν θα ήθελα να είχαμε. Negotiations are what they are. You need to make concessions in order to get concessions. Uh, all in all, I think that we are... Καλά τα πάμε πάντως γενικώς με τα θέματα που είναι υπό επεξεργασία. Είμαστε συνεπείς, έχουμε συνεπιστάσει και θέλω να ευχαριστήσω τους εισηγητές. Προείδερευσα όλων των τιμένων διαλόγων. Αλλά βέβαια η ευθύνη για την ενέργεια των διαπραγματεύσεων να απόκειται στις αντιπροσωπείες του Κοινοβουλίου και βέβαια στους εισηγητές τους εκάστοτε. Παρατηρήσεις υπάρχουν. Εγώ λοιπόν σας λέω διαβάστε αυτές τις εκθέσεις. Σημείο 20, δραστηριότητες εποπτικών ομάδων. Κίνα. Είναι εδώ Χέλμουτ Σόλτς. Μπορείς το να μας κάνεις μια σύντομη παρουσίαση. Να μας ενημερώσει την κατάσταση. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είχαμε την ένατη συνεδρία αυτής της εποπτικής ομάδας. Και η ΓΑΜΑ Εμπόρ κλήθηκε να μας ενημερώσει για την κατάσταση σε σχέση με το άνοιγμα του πρώτου γύρου διαπραγματεύσεων για την επενδυτική συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση ε, Κίνα. Και για μια ακόμη φορά τονίστηκε ότι το βασικό ενδιαφέρον τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τα επενδυτικά να σχετίζονται με την πρόσβαση στις κινέζικες αγορές. Η κινέζικη πλευρά έδειξε κάποιο ενδιαφέρον να το αντιμετωπίσει αυτό το θέμα, αλλά με αντάλλαγμα μερικοί θέλουν περισσότερα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόθεση των συμφερόντων των κινέζικων εταιριών στις ευρωπαϊκές αγορές. Σημαντικό αυτό το σημείο. Δεύτερον, είχαμε μια ευρύτερη συζήτηση για τις προσδοκίες και το πολιτικό πλαίσιο. Για μια ακόμη φορά τονίστηκε ότι με την τρίτη συνεδρίαση για τις Επιτροπές Κομμουνιστικού Κόμματος, εκεί τονίστηκε ότι είναι σημαντικό να υπάρξει μεγαλύτερη οικονομική συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και να υπάρξει εμβάθυνση στις μεταρρυθμίσεις ώστε να γίνουν οι Κινέζοι ένας πιθανός εταίρος μεταξύ των εμπορικών δυνάμεων Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων. Δηλαδή, οι Κινέζοι καταλαβαίνουν ότι η διμερή συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση θα συμβάλλει στην ε, δυνατότητα εκείνα να γίνει δυνητικά ένας ε, σημαντικός εταίρος μέσα στο πολυμερές εμπορικό σύστημα στο πλευρό άλλων σημαντικών χωρών. Και να σας πω ολοκληρώνοντας ότι ομάδα, στην εποπτική ομάδα ε, προσωπήθηκαν όλες οι πολιτικές ομάδες. Πράγματι είναι πολύ σημαντική αυτές οι διαπραγματεύσεις και γιατί είναι η πρώτη επενδυτική συμφωνία που διαπραγματευόμαστε και γιατί δεν διαπραγματευόμαστε με την Κίνα και δεν υπάρχει ισότιμο πεδίο σε ό,τι αφορά την πρόσβαση της ε, Κίνας σε στην Ένωση. Ελλάδα, Πορτογαλία. Να σας αναφέρω παράδειγμα. Και τη δική μας πρόσβαση στην Κίνα. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με αυτέ τι διαπραγματεύσει. Κολομβία, Περού, δεν είναι εδώ ο κύριο Ντάβιντ. Ούτε ο κύριο Λάγκεν είναι εδώ όμω. Ο κύριο Κούτα, μήπω. Α, για το Μερκοσούρ. Λοιπόν, για την Κολομβία και το Περού συνεδρίασε η υποπτική ομάδα με εκπροσώπους των δύο αυτοχωρών, τους πρέσβεις, την κυρία Ρονκίγιο και τον κύριο Ριμπέρα για την κατάσταση, που έχει, ε, την κατάσταση των, ε, της εφαρμογής των συμφωνιών με τις χώρες αυτές. Το ίδιο θα γίνει το Μάρτιο στο Λόκου. Θέλω να σας πω ότι οι συμφωνίες αυτές ήταν οι πρώτες που αποφάσισαν τα κοινοβούλια να ζητήσουν οδικό χάρτη από τους εταίρους για θέματα εργασιακά και μετά να δοθεί συνένεση και έγκριση. Άρα δεν πρέπει μόνο να παρακολουθούμε την ε, συμφωνία αυτή, αλλά και τον οδικό χάρτη για τις προϋποθέσεις οι οποίες ε, αναφέρονται σε επίσημα έγγραφα το οποίο έκριναν και οι δύο χώρες. Έχουν δηλαδή αναλάβει δεσμεύσεις άμεσα προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και όχι μόνο προς την Ένωση γενικά. Αυτό είναι σημαντικό. Δεν είναι ένα χαρτί απλό δηλαδή. Πρέπει πραγματικά να εκπληρώσουν αυτές οι δύο χώρες τις δεσμεύσεις τους, γι' αυτό και θεωρώ ότι η αντιπροσωπεία μας είναι πολύ σημαντική. Εκουαδόρ Χέλμουντ Σόλτς. Είχαμε την πέμπτη συνεδρία της εποπτικής ομάδας αυτή την εβδομάδα. Πάλι μας ενημέρωσε το ΓΔ Εμπόριο για την εστίαση, το επίκεντρο των διαπραγματεύσεων. Δεν πρόκειται για ένα πλήρη γύρο διαπραγματεύσεων, αλλά για πιθανές προσαρμογές ορισμένων κεφαλαίων της πολυμερούς αυτής συμφωνίας, της πλειονομερούς μάλλον συμφωνίας με Κολομβία, Περού και ίσως και άλλες χώρες το Εκουαδόρ, ο το Δεκέμβριο αποφάσισε να ανανεώσει τις διαπραγματεύσεις, συνεχίσει. Πρώτη έγινε στα μέσα Ιανουαρίου. Τέσσερις ομάδες εργασίας είχαμε για πρόσβαση αγοράς, υπηρεσίες, δημόσιες συμβάσεις και γεωγραφικές ενδείξεις. Ήταν μια ενδιαφέρουσα ευρύ ανταλλαγή απόψεων. Ρωτήσαμε και για άλλες επιπτώσεις, ε, τον αντίκτυπο των συμφωνιών γενικώ στην οικονομική πραγματικότητα του σημερινού και τι <clears throat> συνεπάγεται και για τις άλλες χώρες. Εισαγωγές, εξαγωγές μπανάνας, εμπλέκονται για χώρες της Ένωσης. Για το βιομηχανικό τομέα επίση ρωτήσαμε ποια ανταλλαγή, ποιον προϊόντων ανταλλαγή θα μπορούσε να υπάρχει. Μετά από αυτή την ανταλλαγή απόψεων, τονίσαμε ότι θα πρέπει πολύ σύντομα να γνωρίζουμε τι θα γίνει με το δεύτερο γύρο. Δεν υπάρχει ακόμη ημερομηνία. Δηλαδή να συγκληθεί δεύτερος γύρος αυτή την εποπτική ομάδα ή να δοθούν συστάσεις στο νέο κοινοβούλιο για να συνεχίσει αυτό το έργο. Και από κοινωνική και οικολογική πλευρά ή πλευρά ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι σημαντικέ οι διαπραγματεύσει αυτέ. Τι θα είναι, μια, μια τυπική συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών ή κάτι αντίστοιχο με αυτό, με την κολλήμη και το ΠΕΠ. Ήταν σαφή η Πρέπει να προσχωρήσει στην εφιστάμενη συνθήκη ο σημερινό Πρόεδρος, και εγώ φυσικά και υποστηρίζω την Κομισιόν, Σόλτς. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι θα είναι εύκολες οι διαπραγματεύσεις. Γιατί υπάρχουν οι λόγοι του οποίου έφυγαν το 2009. Οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα. Και όλα αυτά περιορίζουν κάπως τα περιθωρία λιγμών ε, των ε, της πλευράς του σημερινού στις διαπραγματεύσεις. Ως εισηγητής για τις εμπορικές σχέσεις θα έλεγα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτική και να εξετάσει ε, πολύ προσεκτικά τι ζητά και τι προσφέρει. Για να δούμε πού μπορούμε να είμαστε στο δυνατόν πιο ευέλικτοι. Για να αντιμετωπίσουμε με την κατάσταση. Πρώτα, ευχαριστώ Χέλμ. Το Μέρκοσούρ είναι το επόμενο θέμα. Ο κύριος Κούτας Τίποτα καλό νέο υπάρχει. Πρόεδρε, δεν μπορώ να πω αν ή αρνητικά τα νέα, αλλά πρέπει να γνωρίζετε ότι ναι, διαπραγματευόμαστε εδώ και 15 χρόνια. Έχουμε προγραμματίσει αυτή την ομάδα παρακολούθηση γιατί αναμέναμε να υπάρξει ανταλλαγή ε, απόψεων του τελευταίου μήνε του περασμένου χρόνου, το Δεκέμβριο. Δυστυχώ αυτό δεν συνέβη σύμφωνα με τα τελευταία νέα, διότι χτε και σήμερα τα μέλη του Μερκοσούρ ε, συσκέπτονται στο Καράκας αποφάσισαν να θα μας ενημερώσουν, ε, δεν ξέρουμε όμως πότε. Άλλο πρόβλημα είναι η επερχόμενη ε, αλλαγή προεδρίας της Μερκοσούρου που θα έπρεπε καταρχήν να είναι η Αργεντινή, ε, αλλά η Αργεντινή έχει προβλήματα όσον αφορά αυτή την ανταλλαγή ε, προσφορών. Ε, Πάντω ελπίζω και όπω κατά μας είπε και ο κύριος και από την ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ Εμπορίου, εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση είμαστε έτοιμοι να κάνουμε ανταλλαγή και ελπίζουμε ότι θα έχουμε εταίρο σε αυτή την ανταλλαγή. Θα δούμε αν θα γίνει το Μάρτιο. Και άλλη μια πληροφορία που νομίζω είναι σημαντική. Στη διάρκεια των μηνών αυτών, στα τέλη Φεβρουαρίου, θα έχουμε και μια διάσκεψη κορυφής Ένωση Βραζιλία και θα μπορούσαμε ίσως, και να το συζητήσουμε. Η Βραζιλία, η Ουρουγουάη και η Παραγουάη θα μπορούσαν να αποκοπούν και να αφήσουν Αργεντινή πίσω. Να υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Η Κομισιόν είπε ότι το περιμένει αυτό, αν η Αργεντινή δεν μπορέσει να μπει σε αυτή την ανταλλαγή προσφορών. Ταϊλάνδη τώρα, ο Ντέιβιτ Μάρτιν. Ο Φρανκ Ρούζ είναι ο εισηγητής, αλλά δεν μπορούσε να είναι σήμερα παρόν, οπότε σα ενημερώνω. Η Κομισιόν μα ενημέρωσε για τον τρίτο γύρο διαπραγματεύσεων, Όπω θα γνωρίζετε η πολιτική κατάσταση στην Ταλάνδη είναι εξαιρετικά δύσκολη αυτή τη στιγμή. Ε, από όσο γνωρίζω, ο επικεφαλή διαπραγματεύτη δεν μπορεί να είναι παρόν λόγω τη κατάσταση, αλλά έχει σημειωθεί πρόοδο για θέματα όπω ε, κανόνε προέλευση, ε, διευκόλυνση εμπορίου, αλλά και κάποια μη επίμαχα θέματα. Αλλά τα μεγάλα επίμαχα θέματα όπως ο τόνος, ε, φαρμακοβιομηχανία κτλ. δεν συζητήθηκαν. Και μάλιστα δεν ορίστηκε και ημερομηνία για τον τέταρτο γύρο. Τουλάχιστον μέχρι την τελευταία φορά που ενημερώθηκα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τους ε, Ταϊλανδούς γιατί εποφελούνται από τις γενικευμένες προτιμήσεις που εκπνέουν όμως το 2015. Δεύτερο τμήμα της συνάντησης αφορούσε το γιατρούς χωρίς σύνορα και την φαρμακοβιομηχανία για τις ευρεσιτεχνίες και την προστασία αυτών μέσα στο πλαίσιο της ε, Συμφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών. Και μας αποκάλυψαν ότι είναι πολύ δύσκολο για την Κομισιόν να βρει μια διατύπωση που θα λέει πρόσβαση ναι μεν στα φάρμακα αλλά θα δίνεται και στην ε, φαρμακοβιομηχανία ε, μια αποζημίωση για τις επενδύσεις. Ναι, η Ταλάβη περνά πολύ δύσκολες πολιτικές στιγμές. Είπα Είμαι εγώ ο μόνιμος εισηγητής. Έγιναν ε, ένα σωρό συναντήσεις. Τελευταία 22 Ιανουαρίου με τον την τότε αναπληρώτρια ESPR Μίριαμ Σαπίρο, που, που έφυγε απεχώρησε από τη θέση της μετά από μια-δύο μέρες αλλά ήταν υπεύθυνη για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Και γνώριζε πάρα πολύ καλά τα θέματα από πλευράς ε, των ΙΠΑ. Είχαμε λοιπόν μια πολύ ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψεων, αλλά φυσικά όλα τώρα αυτά οδηγούν στη συνάντηση ψηλού επίπεδου ανάμεσα στον Επίτροπο Ντεγκούχτο και τον ομόλογο του τον είπα για να δουν και να επικυρώσουν τι έχουν κάνει οι διπραγματευτές και να προχωρήσουν. Δεν έχουμε εκπλήξεις εκεί, όλα προχωρούν κατευχήν. Οι προσφορές προετοιμάζονται για την πρόσβαση στην αγορά, τόσο για τα αγαθά όσο και για νομικούς φραγμούς για τις υπηρεσίες και τα αγαθά και ως εκ τούτου θα περιμένουμε για το ανακοινωθέν από τον Φρόμεν και τον Τιγκούχτ την επόμενη εβδομάδα στη Ουάσιγκτον. Να έχετε το νου σας, ε, λοιπόν, στην ε, γάμα δέλτα εμπορίου. Εγώ είμαι αισιόδοξο για το αποτέλεσμα. Μπορεί δηλαδή οι διαπραγματευτές να πάρουν μια πιο ισχυρή εντολή για να κινηθούν. Εν τω μεταξύ, όπω γνωρίζετε, η Κομισιόν αποφάσισε να κάνει μια διαβούλευση για τμήμα της, ε, του κεφαλαίου των επενδύσεων, δηλαδή για τους μηχανισμούς ε, προστασίας των επενδύσεων ώστε να καταλήγουν περισσότερο σε διατησία και όχι στο δικαστήριο. Αυτό έγινε επίμαχο θέμα. Η Κομισιόν ξεκίνησε διαβούλευση. Θα υπάρξει κάποιο κείμενο ολοκληρωμένο γι' αυτό το κομμάτι αυτού του κεφαλαίου. Και εδώ διαβούλευση σημαίνει όχι μόνο το κοινό αλλά και τα κρατημέλη και νομίζω πως είναι μια εξαίρετη ευκαιρία για τα κρατημέλη να πούνε στα θεσμικά όργανα, δηλαδή στην Κομισιόν, το Συμβούλιο και εμάς εδώ στο Κοινοβούλιο, ποια είναι η θέση τους ε, σε σχέση με την ISDS. Βιετνάμ. Δεν έχουμε εδώ κανέναν εισηγητή. Έχω εδώ ένα σημείωμα. Η ε, ομάδα παρακολούθησης έκανε μια, η υποπτική ομάδα έκανε μια συναδρίαση στις 31 ε, Ιανουαρίου για να ανταλλάξει απόψεις για τον έκτο γύρο διαπραγματεύσεων και για τις διαπραγματεύσεις για τον έβδομο γύρο. Σύμφωνα με τις πηγές μου, τα πράγματα προχωρούν ομαλά Υπάρχει πρόοδος λοιπόν και μάλλον θα ολοκληρωθούν πριν από το τέλος. Τέλος Μαγκρέμπ. Η συγκίτρινη και η Μαρία Σαρνέζ έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε ολοκληρώνεται η συμφωνία, η συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών. Έγιναν τρει γύροι και ένα τέταρτο γύρος θα γίνει φέτο. Εμείς συγκεντρώσαμε την ομάδα παρακολούθησης τρει φορές. Μαζί με τον David Μάρτιν μάλιστα κάναμε Μασρέκ και Μαγκρέμπ. Η τελευταία μας συνεδρίαση έγινε το Δεκέμβριο και αφιερώθηκε σχεδόν αποκλειστικά στην εφαρμογή της Γεωργικής Συμφωνίας και στο θέμα των γεωγραφικών ενδείξεων. Είχαμε τη ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ Άγκρη που ήταν παρούσα, μας ενημέρωσε για όλα. Όλα πάνε πάρα πολύ καλά, έχει δημοσιευθεί και ένας κατάλογος. Βλέπουμε προφανώς ότι δεν είναι στο ίδιο επίπεδο. Για παράδειγμα, εμείς θα προστατεύσουμε, θα υπάρχει γεωγραφική ένδειξη 16-20 έναντι 3020 για την Ένωση ε, ενώ είναι 16-20 για το Μαρόκο, δεν απειλούμεθα. Και έπειτα κάτι ακόμα, έχουμε το λάδι... Ε, το λάδι αργάν που είναι ε, κατεξοχήν προϊόν του Μαρόκου ε, και θέλει να το προστατεύσει. Το Μαρόκο θέλει να εγγραφούν ειδικέ του γεωγραφικέ ενδείξει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να μπορεί να χαίρει των μπλε και πράσινων λογοτύπων ε, τη Ευρωπαϊκή Ένωση για τι γεωγραφικέ ενδείξει. Εγώ θα ήθελα να το δούμε αυτό το θέμα πριν να το διώξουμε και να επανέλθουμε να δούμε μήπως μπορούμε να είμαστε ανοιχτοί εδώ. Πιστεύω πως πρέπει να το σκεφτούμε. Τι υπάρχει ήδη, υπάρχουν ήδη αντιδράσεις από πλευρά τη Κομισιόν. Ε, όχι, η Κομισιόν δεν τα πέριψε. Του ζητήσαμε να το σκεφτούν. Δεν έχω ακόμα ακούσει κάτι νεότερο. Τώρα, ένα σημείο το οποίο βεβαίως είναι πάντοτε ευαίσθητο, αλλά δεν έχουμε πρόβλημα εκεί, Ωστόσο, είναι το θέμα της Δυτικής Σαχάρας, όπου οι γεωγραφική ενδείξεις συνδέονται με, την, με το, το, την εδαφικότητα, το έδαφος, και εκεί δεν υπάρχει καμία γεωγραφική ένδειξη για την ώρα, για τη Δυτική Σαχάρα, την επικράτη της Δυτικής Σαχάρας. Αυτά λοιπόν, όλα πάνε πολύ καλά και στη Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών και για το θέμα των γεωγραφικών ενδείξεων. Συνάδελφοι, καλύψαμε ε, τα θέματα όπου είχαμε εποπτικές ομάδες και διερωτάμε αν καλύψαμε και όλες τις ε, διαπραγματεύσεις με όλες μας τις εποπτικές ομάδες. Ήταν εξαιρετική ιδέα το να φτιάξουμε αυτές τις ομάδες. Να ευχαριστήσω δε τους εισηγητές όλους που ήταν ε, οι εμψυχωτές αυτών των ομάδων και συνέλεξαν πληροφορίες, απόψεις, ε, συμμετείχαν σε συζητήσεις με τρίτα μέρη, γιατί διαφορετικά αυτό δεν θα είχε γίνει, δεν θα είχε καταστεί δυνατό. Είναι τόσο ευρία τα θέματα που δεν θα μπορούσαμε να τα έχουμε καλύψει με τις τακτικές συνεδριάσεις της Επιτροπής μας και βέβαια αυτό αποτελεί τιμή και για την Κομισιόν που ασκεί πολύ φιλόδοξη εμπορική πολιτική. Εν γέννη πάντως τα πράγματα πάνε καλά και αυτό είναι καλό για ολόκληρη την Ένωση. Αν όλα πήγαιναν τόσο καλά όπως στην εμπορική πολιτική, η Ένωσή μας θα ήταν σε πολύ καλύτερη φόρμα από ό,τι είναι αυτή τη στιγμή. Σας ευχαριστώ πολύ όλους. Δεν έχουμε τίποτα στα διάφορα. Η επόμενη μας συνεδρίαση προβλέπεται στις 19 και 20 Μαρτίου.